Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση λοιπόν. Το πρακτικό της χρησινής συνεδριάσεως έχει ήδη διανεμηθεί. Ερωτώ εάν έχετε ενστάσεις. Όχι. Καλώς λοιπόν εγκρίνεται το